Αναρχίζει λοιπόν η συνεδρίαση η οποία είχε διακοπεί στην προηγούμενη, στο τέλος της προηγούμενης Ολομέλειας. Τα πρακτικά ε, της προηγούμενης συνόδου της, 15, 5ης Μαΐου του 2011 ε, περιέχονται ήδη στο φάκελό σας. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις τα πρακτικά εγκρίνονται.